Κυρίες και κύριοι, μεγάλη τιμή που κηρύσω την έναρξη των εργασιών της ομάδας εργασίας μας. Σήμερα θα συζητήσουμε την Ευρώπη της δικαιοσύνης, ε, την αύξηση του δημοκρατικού ελέγχου και της ασφάλειας δικαίου σε εθνικό επίπεδο, τοπικό επίπεδο αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρετίζω τον αντιπρόεδρό μου, τον κύριο Μέντες Δεβίγο. Και επίσης τον κύριο Αυσάν που είναι συγητής του σημερινού μας θέματος, Έλενα Γκαϊντούσκοβα από τη γερουσία του, της Τεχικής Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δική μου, να σας συστηθώ δηλαδή. Θα ήθελα να σας αναφέρω εν συντομία πώς ε, θα προχωρήσουν οι εργασίες μας. Η συζήτηση θα διέπεται από τους ίδιους κανόνες όπως ισχύει και στην Ολομέλεια. Πρώτα απ' όλα δηλαδή θα μιλήσουν δύο μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων και μετά θα μιλήσει ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη σειρά με την οποία θα έχετε ζητήσει το λόγο. Όταν σηκώνετε την πορτοκαλί σελίδα σας, το πορτοκαλί φίλο. Η γραμματεία θα είναι υπεύθυνη για την κατάτηση του καταλόγου των αγορητών. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Όπως και στην Ολομέλεια, θα έχετε περίπου τρία λεπτά στη διάθεσή σας για τις παρεμβάσεις σας. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Αυσάν, Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Να μιλήσω λίγο για το θέμα συζήτησής μας σήμερα στην ομάδα εργασίας μας. Όπως όλοι γνωρίζουν υπάρχει ένας γενικότερος στόχος να επιτύχουμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης όπου θα λειτουργούν αρμονικά και αποτελεσματικά όλα τα ένομα συστήματα των ε, κρατών μελών. Σεβόμενοι πάντοτε τις εθνικές νομικές παραδόσεις. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση του χώρου δικαιοσύνης είναι η ενίσχυση συνεργασία για την βία αναγνώριση των αποφάσεων, των δικαστικών αποφάσεων. Αυτό απαιτεί την κατάλυση όλων των φραγμών που υπολείπονται μια ευρεία αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων συνεπάγεται ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν εμπιστοσύνη στα ένομα στήματα των λοιπών κρατών μελών και στις αποφάσεις τους, τόσο ώστε να διεξάγεται η διαδικασία του εκτελεστού τίτλου στον τομέα του ε, αστικού δικαίου. Αν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να διευρυνθεί αμοιβαία αναγνώριση και σε άλλους τομείς. Γαμικές σχέσεις, διαθήκες, ε, κληρονομιές. Στα πλαίσια αυτής της ε, συνεργασίας ε, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για την αναγνώριση των αποφάσεων, αλλά πρόκειται να γίνουν και άλλα πολύ σημαντικά βήματα ε, μιλάμε για πολλά διαφορετικά στάδια της ποινική διαδικασίας και πολλές και διαφορετικές ε, αποφάσεις. Κυρίως πρόκειται για διοικητικές αποφάσεις, προστασία των θυμάτων, εγκληματικών πράξεων, απώλεια των προσωπικών ε, δικαιωμάτων και έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες διότι πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει διάφορα μέτρα ε, προς όλους τους, ε, που, ε, τους λειτουργούς στον δικαστικό τομέα των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε κοινά πρότυπα, χρειάζεται προσέγγιση ανάμεσα στις εθνικές νομοθεσίες για κάποια ζητήματα του ποινικού δικαίου που ήδη έχει αρχίσει και πρέπει να συνεχίσει και κυρίως πρόκειται για διασυνοριακές σοβαρές εγκληματικές πράξεις, τρομοκρατία, οργανωμένη εγκληματικότητα και εγκλήματα που πλήττουν βασικά ζωτικά οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών. Ε, τα γενικά πρότυπα θα ε, αναπτυχθούν περιττέρω και θα υπάρξει ευρύτερη αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων. Για το αστικό δίκαιο θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο νέα προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών διαμέσου των ελαχίστων κοινών προτύπων. Και πέρα από την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και τα κοινά πρότυπα, θα πρέπει να επιδιώξουμε την διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των πολιτών, ε, μιλώντας για το ευεργέτημα της παινίας ή η βοήθεια με την γλώσσα ε, στα πλαίσια δικαστικής ε, διαδικασίας και υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε όλος ιδιαίτερως για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Πρώτον, Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων δεύτερον. Πώς ε, μπορούμε να ενισχύσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τρίτον, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη. Αναμένω να γίνει μια καρποφόρα και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αυσάν. Εκπρόσωπε του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Και τώρα, μετά την εισαγωγή του εισηγητού, να δώσω στον Στάνισλαβ Σαρκότσκι από την ε, γερουσία της Πολωνίας το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Είμαι από μια χώρα που δεν θεωρείται πάντα δεδομένη αυτή η κατάσταση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν οι πολίτες μας σε μια χώρα όπου βασική αρχή που επικρατεί είναι το κράτος δικαίου και οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι προβλέψιμες και εφαρμόζονται σύμφωνα με τον νόμο και είναι υπεύθυνε όλο και περισσότερο οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πόσο καλό κάνει η Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Δεν αφορά μόνο τα ταξίδια και την παιδεία, αλλά και, και το επιχειρήν. Ε, κινούνται επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και η παγκοσμιοποίηση, η πρόσβαση στο διαδίκτυο σχεδόν υποχρεώνουν τις εταιρείε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε, όλες, σε πολλές χώρες. Το πρόγραμμα τη Στοκχόλμης αναφέρεται στην Ευρώπη της δικαιοσύνης. Έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνους ε, που έχουν τις επιχειρήσεις και δικούν τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό της κοινή αγοράς και να εφαρμόσουμε τις συνθήκες. Και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να καταργήσουμε, να άρουμε μάλλον τα εμπόδια που υπάρχουν όσον αφορά την αναγνώριση όλων των νομικών πράξεων σε όλα τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε σχέσεις και με τις τρίτες χώρες. Έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα των πολιτών μας λαμβάνονται υπόψη. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πρώτερες διμερείς σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των τρίτων χωρών. Θέλουμε να έχουμε μια συνεκτική κοινή πολιτική σε αυτό το τομέα, αλλά θα πρέπει να βρούμε και τη σωστή ισορροπία, ώστε τα εθνικά συμφέροντα να λαμβάνονται υπόψη. Υποστηρίζω ολόθερμα την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων. Είναι βάση της συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να σεβόμαστε και τις διάφορες νομικές παραδόσεις των κρατών μελών. Και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πω ότι έχω αμφιβολίες κατά πόσο αυτός ο κανόνας περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως θα πρέπει να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει και διοικητικές αποφάσεις. Αυτή η αρχή αναπτύχθηκε, δημιουργήθηκε για δικαστική συνεργασία και υποθέτουμε ότι θα τηρηθούν ψηλότερες προδιαγραφές. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε διοικητικές υποθέσεις ε, είναι πιο αυτόματες όσον αφορά την εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση είναι πολύ πιο παρακινδυνευμένη. Αν θέλουμε να καταργήσουμε την διαδικασία εξεκουάτορ σε άλλους τομείς που, που καλύπτονται από νομοθεσία της κοινότητας, αυτό σημαίνει ότι το δικαστικό σύστημα ε, θα λειτουργεί πιο όμαλα τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν θέλουμε το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να συλλέξουμε τις εμπειρίες μας, να τις ανταλλάξουμε, να τις συζητήσουμε, θα πρέπει, θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών επίσης στην κοινότητα. Το πιο σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη πρέπει να έχουμε ένα στον άλλον και αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση για όλους μας. Ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, θεσπίζουμε τον νόμο που μετά εφαρμόζεται. Και είναι τεράστια πρόκληση αυτή για τους πολιτικούς. Θα ήθελα να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Νομίζω ότι μπορούμε να αποδείξουμε ότι εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και αυτό θα είναι ένα υπέροχο μήνυμα θα μπορούσαμε να στείλουμε στους πολίτες μας. Θα καταλάβουν ότι παντού επικρατούν οι ίδιοι όροι και τηρούνται οι ίδιες, πληρούνται οι ίδιες προδιαγραφές. Θα ήθελα να ζητήσω από τους όλους, από τους όλους τους να τηρήσουν το χρονικό τους όριο από την Ιταλική Γερουσία, ο κ. Μοϊτάτε. Και μετά ο Αντρίου Μπραμς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να πω κάτι περισσότερο από αυτά που κατάφεραν να, πούν, να πω στην, στην Ολομέλεια. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να κινηθεί γρηγορότερα διότι έχουμε μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά ένα πρόγραμμα διοργάνωσης της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Δηλαδή, διοργάνωση για προάσπιση της ελευθερίας όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Για να γίνει αυτό, δεν χρειάζεται πλέον να αναλύουμε το, το εγκληματικό φαινόμενο που κινείται διεθνώς και έχει διεθνείς βάσεις και διευρύνει τη βάση συνεχώς. Δεν χρειάζεται πλέον να επαναλαμβανόμαστε και να επαναλαμβάνουμε τι μπορεί να συμβεί σε μια Ευρώπη που είναι στα χέρια της του οργανωμένου εγκλήματος, που βρίσκεται παντού και πλουτίζει συνέχεια το οργανωμένο έγκλημα. Όλα αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, και είναι κάτι και τα χρήματά τους μολύνουν την οικονομία μας. Πρέπει να κινηθούμε σοβαρά στην πράξη, δηλαδή να δημιουργήσουμε τους θεσμούς που ήδη έχουν ε, εντοπιστεί και έχουμε δοκιμάσει ήδη στις χώρες μας, τα κράτη-μέλη, όπως στη χώρα μας στην Ιταλία, που, που θα αναφερθώ και θα πω κάποια πράγματα, ή κάποια πράγματα που ενετόπισε η Ευρώπη με, μέσω συζητήσεων, μέσω ε, προτάσεων. Λοιπόν, οι κοινέ αυτέ ομάδε ε, τη ε, ποινική δικαστική αστυνομία. Διότι γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο και διεθνέ το έγκλημα. Από πέντε άτομα διαπράθεται ένα έγκλημα στην Νότια Ιταλία, στην Καλαβρία και μετά διώκονται και φτάνουν σε μια, και κινούνται στη Γερμανία και γίνεται μεγάλο εμπόριο κοκαίνης στην ε, Αλβανία, οργανώνεται, συνεχίζεται στην Ιταλία, προετοιμάζεται το προϊόν στην Κολομβία και μετά μπαίνουν τόνοι ποσοτήτων και στην κεντρική και στη Δυτική Ευρώπη. Τέτοιο, τέτοια επίθεση εγκληματική πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με μια διεθνή οργάνωση που απαιτεί μια αστυνομία. Έχουμε την Europol, αλλά είναι εντελώ ανεπαρκής. Οπότε θα πρέπει να ξαναπροσδιορίσουμε και θα πρέπει να δώσουμε προκαθορισμένες εξουσίες. Στο Eurojust, παραδείγματο χάρη, το Eurojust θα πρέπει να μεταφραστεί, να γίνει ένα κέντρο συντονισμού. Ε, θα πρέπει να μαζεύουμε τις γνώσεις. Χρειάζεται να έχουμε βάση δεδομένων με στοιχεία διεθνή, ευρωπαϊκά. Χρειάζεται ε, ένα σημείο συντονισμού, ένα φορέας συντονισμού και να δώσει όθηση στην προσπάθεια. Δεν θέλουμε να στερήσουμε τα κράτη-μέλη από διάφορα προνόμια ή διάφορες εξουσίες ή από κυριαρχία. Πρέπει να εμπλουτίσουμε, να ενισχύσουμε αυτές τις, αυτούς τους φορείς, τους τοπικούς και τους κρατικούς. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε πραγματικά τις καθυστερήσεις και τις καχυποψίες κάποιων ευρωδιστακτικών χωρών. Θα πρέπει να δώσουμε ζωή σε αυτούς τους οργανισμούς, δηλαδή να ενισχύσουμε όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τις χώρες που την απαρτίζουν Eurojust, βάσει δεδομένων, ε, πληροφορική να μπει σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει αυτοί οι φορεί να έχουν τι μεγαλύτερε δυνατέ εξουσίε. Είναι κάτι αναπόφευκτο πιστεύω και δεν μπορούμε να καθυστερούμε πλέον. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε, θα πρέπει να καθορίσουμε τα όρια τη εξουσία. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να καθορίσουμε και τι ευθύνε του. Και δεν είναι δυνατόν να, έχουμε, να σκεφτούμε τέτοιου διεθνεί φορεί λησμόνησα να προσθέσω και μια εισαγγελία, διεθνή εισαγγελία, μια ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα, θα έχει πάντα την αρμοδιότητα να γνωρίζει στοιχεία, πληροφορίε που θα προέρχονται από όλη την Ευρώπη και όμω θα μεταφράζονται πληροφορίε σε, ένα, σε γνώσει υπέρ των διαφόρων εθνικών εισαγγελιών από ένα κεντρικό σημείο. Δεν μπορούμε να ελοπίσουμε φορεί τόσο χρήσιμους, τόσο αποτελεσματικούς που θα πρέπει να είναι ισχυρή χωρίς να υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις σωστής δράσεως, σωστής εκτελέσης των καθήκων τους και σωστής απόδοσης ευθυνών. Αυτή η απόδοση των ευθυνών ε, θα πρέπει ε, να ξεκινά από τα κράτη-μέλη αλλά σε κάποια φάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από κάποιο φορέα που εξαρτάται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, ο Άντριου Μπρόμς. Ευρωβουλευτής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις ότι αντίληψη ότι χρειάζεται ένα κοινό εμπορικό σύστημα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δεν είναι ισχύει, γιατί ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ξεχωριστό νομικό σύστημα και για παράδειγμα στο σημαντικό δίκαιο, στην περίπτωση του, του δικαίου κληρονομιάς, εξαρτάται από το τόπο κατοικία και την ε, ηθαγένεια του ατόμου. Ένα έγγραφο το οποίο κυκλοφόρησε από τρεις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπονόησε ότι χρειάζεται ενιαίο συμβατικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Θεωρώ ότι το αγγλικό σύστημα για το συμβατικό δίκαιο έχει αναπτυχθεί συστηματικά και συγκεκριμένα τα τελευταία 400 χρόνια σε ό,τι αφορά το συμβατικό δίκαιο και η ιδέα ότι θα αντικατασταθεί το σύστημα αυτό από ένα ενιαίο κωδικοποιημένο σύστημα θα προκαλούσε φρίκη στους πολίτες μας. Στο ίδιο έγγραφο υπονοείται ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα κοινό νομικό ποινικό σύστημα. Αυτό τι θα σήμαινε ότι θα καταργούταν το δικό μας σύστημα, το οποίο όχι μόνο οδηγεί σε συγκεκριμένα συστήματα, αλλά και αυξάνει τη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά την απόδοση της δικαιοσύνης. Το, το Βρετανικό σύστημα, μάλλον οι Βρετανοί πολίτες θα έφρυταν αν ε, προχωρούσαν αυτές οι δύο δράσεις. Δεν πιστεύω ότι ο κοινός εμπορικός χώρος χρειάζεται να καταπατήσει την εθνική κυριαρχία και την κυριαρχία των νομικών συστημάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σλόπνικ από το Σλοβανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Η δημοκρατία της Σλοβενίας προγραμματίζει το επόμενο πολιτές του πολιτές της πρόγραμμα για το περιοδο 2010-2014 σε ό,τι αφορά το τομέα της δικαιοσύνης. Τα πρώτα βήματα έγιναν κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής και Σλοβενικής Προεδρίας στο πλαίσιο της ομάδας Futura, όπου και συζητήσαμε τους διάφορους στόχους μας σε ό,τι αφορά τον χώρο της ασφάλειας της δικαιοσύνης. Οι προετοιμασίες είχαν ως αποτέλεσμα το έγγραφο του Πρωτορός, το οποίο περιλαμβάνει κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον, για την πιο αποτελεσματική ε, προστασία στον τομέα της δικαιοσύνης, η οποία προαπαιτεί αμοιβαία αναγνώριση. Το δικαστήριο της χώρας προέλευσης θα πρέπει να υπερισχύει και αυτό θα διασφαλίσει την αμοιβαία αξιοπιστία και την ελεύθερη ροή των δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κάποιε βασικέ αρχέ οι οποίε θα ισχύουν. Όπω για παράδειγμα το δικαίωμα των ένομων μέσων τη μερική εναρμόνιση των δικαστικών αποφάσεων σε ό,τι αφορά τις οικονομικές και αστικές υποθέσεις θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταργήσουμε τη διαδικασία εκτελεστού τίτλου, εξεκβάτορ ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία η οποία ε, αποκλείει τη λήψη δικαστικής απόφασης σε άλλη χώρα. Λόγω βασικών διαφορών επί της αρχής μεταξύ των ε, δικαστικών συστημάτων των χωρών θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί στην προσέγγιση μας. Θα πρέπει να δράσουμε με συνεκτικό τρόπο, να σεβαστούμε τις αρχές της ε, επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαδικασίες για την αμοιβαία αξιοπιστία, όπως για παράδειγμα τα βελτιωμένα σχετικά πρότυπα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα της ε, διερμηνίας. Η Δημοκρατία της Σλοβενίας υποστηρίζει τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου για τα δικαιώματα περί διερμηνίας, με κάποιες ίσονο σημασίας ε, τροποποίησης. σε ό,τι αφορά την μετεκπαίδευση των χρηστών και την, ε, τις ποινικέ διαδικασίες, όπως για παράδειγμα στα πλαίσια της Eurojust, ε, πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία. Επιπλέον, η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα δικαστικά συστήματα άλλων χωρών είναι επίσης πολύ σημαντική, γιατί αυτό θα καταλήξει τελικά στην ε, οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σλόπνικ. Επόμενος. Ο, Λόρδο Λόρδος Από τη Βουλή των Λόρδων και ο Γιούλας Σαμπατάουσκας από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να συνεχίζετε να ζητάτε το λόγο, είτε να ζητάτε άμεσα το λόγο, είτε γραπτό να ζητάτε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να με συγχωρείτε που παραμένω Καθεστώ, διότι πιστεύω ότι εδώ είναι ομάδα εργασία και ίσω είναι πιο εύκολο να εργαστούμε καθήμενοι. Ε, ελπίζω η υποστήριξή μου για την έννοια μιας, ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνη ασφάλεια και ελευθερία, ε, να θεωρηθεί ότι δεν προδικάζει όσα θα ακολουθήσουν. Δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι απλώς ένα εμπορικό σχήμα εμπορικών συναλλαγών. Ε, προσπαθούμε να πετύχουμε πράγματα μέσω του προγράμματος της Τοχόλμης, αξιοθαύμαστα, αλλά όπως προανέφερα σήμερα στην Ολομέλεια, πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να έχει κάποιες προτεραιότητες και στην ομάδα εργασία μας θα πρέπει να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν για να προστατευτούν τα δικαιώματα των πολιτών και να αυξηθούν τα δικαιώματα των πολιτών στην Ευρώπη. Κάποια στοιχεία αναφέρθηκαν ήδη το απόγευμα. Η κατάργηση του εξεκουάτου. Η Επιτροπή μου το υποστηρίζει πλήρως. Ε, είναι πρακτικό όφελος προ εκείνου που ήθελαν ε, να καταφύγουν σε ένδικα μέσα διασυνοριακά και για τις, ε, θα πρέπει στις ποινικέ δίκες αυτά τα δικαιώματα να καλύπτονται ακριβοδίκαια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα εναρμόνιση, δεν σημαίνει εναρμόνιση του ποινικού δικαίου στις χώρες. Εκεί που αντιμετωπίζουμε δυσκολίες είναι όταν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο εμπεριέχει συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ παρανέφερα δύο παραδείγματα εμείς εδώ ε, κινούμαστε σε αριστολογία και κανόνες διαδοχής παραδείγματος χάρη. Ήδη υπάρχει η σχετική πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν συγκεκριμένα και υπάρχει το πιστοποιητικό αυτό διαδοχής κληρονομιάς θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσους ασχολούνται στο, σε αρμόδιους τομείς, θα ήθελα κάτι μέλη θα ήταν ε, κάτι που θα ήταν ε, πρακτικός θετικό για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα οδηγούσε σε οικονομία. Όμως αν ακολουθήσουμε πλήρως αν θέλουμε να ακολουθήσουμε πλήρως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει 27 διαφορετικές ε, νομικές παραδόσεις και νομολογίες. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το οργάνωμα έγκλημα, ε, παράνομη μετανάστευση, εμπόριο λευκής αρκός κλπ. Αυτά δεν μπορούμε να τα πετύχουμε πολύ γρήγορα. Θέλουμε πρακτικά βήματα να βοηθήσουμε τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή, στη δουλειά τους. Σας έδωσα δύο παραδείγματα, τρία παραδείγματα σας έδωσα και διατείνομαι ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα και αυτή η ομάδα εργασία πιστεύω θα έπρεπε να εξετάζει συγκεκριμένα θέματα και να προτείνει συγκεκριμένε λύσει ε, που θα υποβάλει στην ε, ολομέλεια που θα ακολουθήσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Και τέλος, ο Γιούλιος Σαμπατάουσκας από τη Λιθουανία, σε αυτό το γύρο τελευταίος. Κυρία Πρόεδρε, το πρόγραμμα τονίζει τη σημασία των αμοιβαίων, της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων και υποστηρίζει η Λιθουανία την αναγνώριση των αποφάσεων στα θέματα αστικού δικαίου. Θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι αποφάσεις χωρίς ενδιάμεσα μέσα. Ενδιάμεσα στάδια μάλλον. Και υποστηρίζουμε την κατάργηση του εξεκουάτορ που πολύ συχνά ε, χρησιμοποιείται σε άλλα κράτη-μέλη και εφαρμόζεται για να θετηθούν σε ένα κράτο μέλο αποφάσει που έχουν ληφθεί σε άλλο κράτο μέλο. Λοιπόν, θα πρέπει να θετηθούν κατάλληλοι κανόνε για σύγκρουση δικαίων ε, νόμων τάξεων και θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε θέματα κληρονομία, διαζυγίου και σε συναφή. Η Λιθουανία έχει θετική άποψη όσον αφορά την εφαρμογή της αμοιβαία αναγνώρισης σε διοικητικά ζητήματα και θα πρέπει να εξασφαλίζεται τουλάχιστον σε κάποιες διοικητικέ υποθέσεις η αμοιβαία αναγνώριση. Εφαρμόζοντας λοιπόν τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη και αφαιρώντας τα εμπόδια για την αμοιβαία αναγνώριση θα πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε κάποια μέσα που θα βοηθούν την αμοιβαία αναγνώριση. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και, η, ε, και ο σωστός έλεγχος για τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Και θα πρέπει όταν υπάρχει σύγκρουση ενόμων τάξεων να υπάρχουν λύσεις κυρίως σε εμπορικά και αστικά θέματα, εμπορικές και αστικές υποθέσεις. Ε, εκεί σε αυτά τα θέματα η διατύπωση δεν πρέπει να είναι τόσο συγκεκριμένη διότι ίσως σε κάποιους τομείς δεν θα γίνεται, δεν θα είναι πολύ εύκολη η λύση της σύγκρουσης ενόμων τάξεων. Θα πρέπει να εφαρμόζονται και διάφορες προδιαγραφές όσον αφορά τις αστικές υποθέσεις και την αμοιβαία αναγνώριση. Δεν είναι σίγουρο αν, ε, ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε γενική εναρμόνιση. Θα πρέπει η διατύπωσή μας να είναι πιο ξεκάθαρη. και η προστασία των συμβασιακών σχέσεων. Δεν υποστηρίζουμε εναρμόνιση του συμβατικού δικαίου. Στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος προστατεύονται τα θύματα. Να προστατεύονται με διάφορα μέτρα. Άρση ποινική δίωξης να δίνονται σωστές αποζημιώσεις στα θύματα και το καθεξής. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή διατύπωση αυτών των διατάξεων και να υπάρχει διακριτική ευχαίρεια από πλευράς κρατών μελών, να παρέχεται ένα περιθώριο λιγμό στα κράτη-μέλη και να λαμβάνεται υπόψη και η νομική παράδοση των διαφόρων ε, κρατών μελών, προσπαθώντας να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Σας ευχαριστώ. κύριος Τάντας Σουίφκα ζήτησε το λόγο στο μεταξύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ θέρμα για την ευκαιρία που μας δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις για τη δημιουργία αυτού του κοινού χώρου δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια θεσπέσια ευκαιρία για να υπάρξει ανταλλαγή απόψε ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και συχνά διαπιστώνω ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων σε αυτό το τομέα. Είμαι και η εισηγητής του Κοινοβουλίου για την ε, αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 1 για, το για ζητήματα ενοχικού και αστικού δικαίου. όσα άκουσα σήμερα θα έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη σύνταξη της εκθεσής μου. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις Είμαι πεπισμένος ότι αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από όλα είναι μια δυναμική συνεργασία τόσο ώστε να αποκτήσουμε ένα είδος ε, κοινοτική νομικής ε, κουλτούρας. Μιλήσαμε για διαφορετικά ένομα συστήματα, εθνικά ένομα συστήματα. Και μην ξεχνάτε ότι ο τρόπος λειτουργίας τους διαφέρει πολύ από κράτος σε κράτος και δεν επικρατεί και πλήρης εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αν λοιπόν θέλουμε να τελεσφορήσει αυτό το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, οφείλουμε να κάνουμε μία μεγαλύτερη προσπάθεια. Δεν είναι το πρώτο εγχείρημά μας. Αν θέλουμε να στεφθεί με επιτυχία αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να οικοδομήσουμε μία εμπιστοσύνη. Απευθύνω λοιπόν ένα αίτημα προς εσάς, ε, τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όταν πραγματεύεστε αυτά τα ζητήματα στις χώρες σας, έχετε κατά νου αυτόν τον απότερο στόχο της δημιουργίας ε, ε, κοινοτικής ε, νομικής ε, κουλτούρας ή παράδοσης και δεν είναι μόνο θέμα ποιότητας των αλλαγών αλλά και εφαρμογής των ε, νομοθετημάτων της μεταφοράς του στην εθνική νομοθεσία. Σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις και υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που αργούν πάρα πολύ να μεταφέρουν τις οδηγίες και τους κανονισμούς στην εθνική νομοθεσία. Αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τώρα, ως προς την κατάργηση της αρχής ε, του εκτελεστού τίτλου, με ικανοποιεί που υποστηρίζεται αυτήν τη γραμμή. Χάρη σε αυτό θα διευκολυνθεί η διαδικασία για τους πολίτες και θα επισπευστεί. Επίσης, διάφορες εθνικές κυβερνήσεις ε, ζητούν μεγαλύτερο έλεγχο ε, ως προς την εφαρμογή των κανόνων και θα χρειαστεί να θεσπίσουμε ένα νέο σύστημα ελέγχου. Μην ξεχνάμε τις μεγάλες νομικές διαφορές που υπάρχουν στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δίκαιο το βρετανικό διαφέρει πολύ από ε, τα διάφορα δίκαια που υπάρχουν στη Γυραιά Ήπειρο. Ο στόχος δεν είναι να εξομοιώσουμε όλα τα νομικά συστήματα, απλά να τα εναρμονίσουμε, να τα προσεγγίσουμε. Ορισμένε φορές ε, θα πρέπει να προβλέψουμε κοινή ποινή, κοινή κάθριξη α πούμε, αλλά σε άλλους τομείς ε, όπως στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος, ε, μιλώντας για εξωτερικά σύνορα, παραδείγματος χάρη, για εμπόριο ανθρώπων, εκεί μπορούμε να φανταστούμε μια ομοιόμορφη διαδικασία εμπόριο ναρκωτικών. Εκεί χρειάζεται ταχεία εφαρμογή κοινών λύσεων. Ε, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία στα οποία μπορούμε να βασίσουμε τη συζήτησή μας και αν θυμάμαι καλά πριν από ένα χρόνο ε, κάναμε αυτήν την συζήτηση της ποινικοποίηση των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος ε, έγινε μια πολύ έντονη συζήτηση για την επιβολή ποινών σε διάφορα κράτη-μέλη μάθαμε ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά μέτρα ανάλογα με το κράτος μέλος ε, και άλλα στοιχεία και μην ξεχνάτε ότι τελικά καταλήξαμε σε κάποια συνένεση το αποτέλεσμα το δέχτηκαν όλοι και αυτό το λέω για να καταδείξω ότι αν πραγματικά το θέλουμε μπορούμε να ε, καταλήξουμε σε μια κοινή ε, λύση. Συνεδριάζουμε μόνο άπαξ το χρόνο, οπότε θα σας πρότεινα να ενισχύσουμε τη συνεργασία κάποιων ε, επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να υπομιστούμε αυτή την ευθύνη σύντομα. Θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Εφόσον ε, ο ρόλος μας είναι να νομοθετούμε, ας νομοθετήσουμε. Σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας. Ο κύριος Μέντες Δεβίκα, ο συμπρόεδρος μου, θα... Ο, συμπρόεδρο ε, θα πάρει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα... Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με τον με τον κύριο Τρίφια, το συντονιστή της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ε, ε, όντως είναι αναγκαίο να υπάρχουν τακτικότερες ε, συνεδριάσεις και πάντοτε είναι θετική η διακοινοβουλευτική συνεργασία. Δεδομένου ότι θα τεθεί σε ισχύ σύντομα η συνθήκη της Λισαβόνας και δομές αύξησης ως εκ τούτου των ορμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου νομίζω ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα διαφορετικό ρόλο. Ε, χρειάζεται να ενισχύσουμε αυτή τη διμερή συνεργασία ανάμεσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο και τις, Εθνικές τις Επιτροπές των ε, ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Εδώ και 18 χρόνια συμμετέχω στη συνεδριάση της ΚΟΖΑΚ, αλλά συνήθως συζητάμε, κάνουμε μάλλον γενικές συζητήσεις, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. θα θεσμοθετήσουμε αυτή την διμερή συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ανακοινωθεί αυτήν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Θέλουμε να υπάρχει συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για να βρούμε λύσει σε συγκεκριμένα προβλήματα. Είπε ένα συναδελφό νωρίτερα ότι είμαστε βουλευτές και ο στόχο μα είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των συμπολιτών μα να βρούμε απαντήσει σε, σε προβλήματα και συχνά οι απαντήσεις που έχουμε δεν επαρκούν ε, σε εθνικό επίπεδο. Αυτό ισχύει για διάφορους τομείς, γεωργία, το περιβάλλον και ισχύει φυσικά και για όλα αυτά τα ζητήματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. μπορούμε να μιλάμε μόνο για μια αγορά, αναφέροντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι υπεραγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Οι ιδρυτές της Ένωσης στη δήλωση της 9ης ε, Μαΐου ανέφεραν τους στόχους των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και μην ξεχνάτε ότι χάρη στην πτώση του τείχους του Βερολίνου μπορούμε να προάγουμε μια πραγματική πολιτική. Δεν θέλουμε να περιοριστούμε στην ενιαία αγορά ή στο κοινό νόμισμα. Δεν είναι εύκολο βέβαια. Και βλέπετε τι συμβαίνει όταν μιλάμε για την ΚΕΠΑ. Ε, έχουμε κάνει μόνο τα πρώτα βήματα στον τομέα της δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί εξελίξεις. Και θα δούμε σε τι θα μας προσφέρει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Το προηγούμενο πρόγραμμα της Χάγης νομίζω δεν ήταν το καταλληλότερο και δεν σημειώθηκε αρκετή πρόοδος. Όλα είναι ε, ζήτημα συγκυριών. Ε, πρέπει να δούμε τι κινητήρα θα έχει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ξέρετε, κάποια αυτοκίνητα πάνε γρήγορα, αλλά όχι, τι να κάνουμε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ήδη έχουμε καταφέρει να υπογραφεί η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και όπως πολύ σωστά είπατε πρέπει παρά τις επιτυχίες μας να εργαστούμε όλοι σκληρά για να δούμε τελικά, τελικά τι θα εισηγείται το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης. Δεν ξέρουμε τελικά σε ποια συμφωνία θα καταλήξει το Συμβούλιο. Έχω την εντύπωση ότι εάν πραγματικά θέλουμε να δείξουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει μια προστιθέμενη αξία για τους ε, πολίτες, ε, θα το καταφέρουμε. Πρόεδρε, δεν θέλω να είναι η σημερινή συζήτηση όπως τελευταία σκηνή του Καζαμπλάνκα, όπου ο Χάμφρεϊ Μπόκαρτ λέει στο ε, ε, εκεί μπροστά στο αστυνομικό τμήμα ότι αυτό θα μπορεί να είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας. Θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσει μια υπέροχη φιλία μέσα από τη σημερινή μας συνεδρία για να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών της Ένωσης και Πρόεδρε ήθελα ήδη να σας συγχαρώ για τον τρόπο που, με τον οποίο υγείστε των συζητήσεων. Μάλιστα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίως για τη φιλοφρόνηση. Θα ήθελε κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Βλέπω, σηκώσατε. Μπορείτε να συστηθείτε. Ευχαριστώ. Είμαι αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Ενικών Υποθέσεων στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να κάνω κάποιε σύντομε παρατηρήσει για το θέμα το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα και είναι πολύ καθοριστικό άλλωστε. Στην Ισπανία σημειώνονται όλο και πιο πολλά εγκλήματα κατά ανηλίκων. Νομίζω ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ποινική προστασία των ανηλίκων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για όλα τα κρατη και θα πρέπει να ε, γίνει ομογενής η προστασία αυτή των ανηλίκων σε όλα τα κράτη-μέλη. Να ενισχύσουμε δηλαδή και την ποινική ευθύνη των γονέων, για παράδειγμα, όχι μόνο την αστική ευθύνη. Θα πρέπει να ρυθμιστούν επίσης ε, οι εθνικές διετάξεις, αναφορικά, για παράδειγμα, με την προστασία της οικογένειας. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό και το γαμικό δίκαιο θα πρέπει να εναρμονιστεί. Ίσως και το νομικό σύστημα για τα διαζύγια και θα πρέπει να ορίσουμε και μία κοινή μεταναστευτική πολιτική και χρειάζεται έντονος έλεγχος από όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι φορά και τη λατρομετανάστευση. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχεδόν ε, με έπεισε ο συμπρόεδρο να πω και κάτι άλλο. Αλλά ο προηγούμενος ομιλητή μίλησε για την εναρμόνιση. Νομίζω ότι με όλο το σεβασμό αυτή τη δυσκολία αντιμετωπίζουμε όταν ε, διαλέγουμε θέματα όπως για παράδειγμα η εναρμόνιση του γαμικού δικαίου και του συμβατικού δικαίου. Φαίνεται ότι καμιά φορά υπάρχει πειρασμός να θεωρήσουμε ότι αυτό θα αποβεί προ όφελο των πολιτών, αλλά δυστυχώ αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα και προηγουμένω. Θέλουμε να βρούμε συγκεκριμένα σημεία που μπορούμε να τράσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε και άλλου τομεί, αλλά στον κατάλογο προτεραιοτήτων θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να πετύχουμε βραχυπρόθεσμα. Και να πω προ έναν συνάδελφο, ο οποίο αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το εξή δεν είμαστε κατά όλου του προγράμματος της Στοκχόλμης. Είμαστε μάλιστα υπέρ του προγράμματος της Στοκχόλμης, αλλά δεν μπορούμε να υποθέτουμε ότι πολλά άλλα ε, σημεία στα οποία θέλουμε να βρούμε κοινό τόπο και τα οποία είναι πολύ χρονοβόρα και δύσκολα να επιτευχθούν και θα προαπαιτούν εναρμόνιση 27 διαφορετικών ενόμων συστημάτων το γεγονός ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει το ξεχωριστό Βρετανικό δίκαιο, δυσκολεύει περισσότερο ακόμα την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε συγκεκριμένες δράσεις, εφικτές, οι οποίες δεν αποτελούν μόνο ε, φιλοδοξίες. Σας ευχαριστώ. Είμαι βέβαιη ότι έχετε δίκιο και βλέπω να ζητά το λόγο και κάποιο άλλο ομιλητή. Παρακαλώ δηλώστε το όνομά σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι που δεύτερο λόγο. Αλλά μιας και έχουμε ώρα μέχρι τις 7 και η ώρα είναι μόλις 6, νομίζω ότι έχουμε λίγη ώρα ακόμα για να συνεχίσουμε τον διάλογο μας. Δεν κατάλαβα από αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι αντίθετο ε, με το Βρετανικό δίκαιο. Όχι, απλά αναφέρθηκα σε διάφορους ευρωσκεπτικιστές που είχαν πάρει το λόγο στην Ολομέλεια και τάχθηκαν κατά των κοινών λύσεων. Αυτό φυσικά δεν με παρεμποδίζει δεν με ενοχλεί. Αντιθέτω, μου δίνει έναυσμα να αναζητήσω περισσότερα σημεία στα οποία μπορούμε να βρούμε μία συμφωνία. Για τον συνάδελφο από την Ισπανία. Η Ισπανική Προεδρία, η οποία θα έρθει, είναι η επερχόμενη, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν συζητήσαμε ωστόσο κάτι πολύ βασικό το ποια θα είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει και όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στα τέλη της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας συζητήθηκε η γνωμοδότησή μου και εγκρίθηκε μάλιστα όπου αναφέρθηκε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούν θα χρειαστεί κάποιος καιρός ακόμα, ίσως όχι πολλά χρόνια, αλλά σίγουρα κάποιος καιρός. Και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη μπορούν να συνάψουν συμφωνίες και με τρίτα κράτη ακόμα και αν το περιεχόμενο των συμφωνιών αυτών ε, εμπίπτει σε αποκλειστικές αρμοδιότητες της κοινότητας. Αυτό καταδεικνύει ότι δεν χρειάζεται η κοινότητα να αποφανθεί για όλους τους τομείς που αφορούν τα 27 κράτη-μέλη για μεμονωμένα ζητήματα τα οποία μπορούν φυσικά να τα πραγματευτούν τα κράτη-μέλη της Ένωσης με τρίτα κράτη. Αυτό είναι κάτι το θεμητό. Όταν υπάρχουν, για παράδειγμα, συγκεκριμένοι γεωγραφικοί όροι, ιστορικές συνθήκες και ούτω καθεξής. Να δοθεί δηλαδή δυνατότητα ε, συνάψης δημερών συμφωνιών ακόμη και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γενική αρμοδιότητα επί του τομέα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή μια ρεαλιστική προσέγγιση, να αναζητήσουμε πραγματικές λύσεις. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή το μελλοντικό κοινωτικό δίκαιο το οποίο ασφαλώς και θα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, θα απολαμβάνει και τις υποστήριξεις των πολιτών της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαριτάτη από την Ιταλία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να καταχραστώ τις υπομονής των συναδέλφων και τη δική σας, αλλά δράτω από αυτή την πληθώρα χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας για να θέσω ένα ερώτημα σε όλους μας και απευθυνόμαστε προς την Προεδρία. Όλοι μας συμφωνούμε όσον αφορά τη δρομολόγηση του νέου συστήματος αυτού συνεργασίας Ακολουθώντα την πορεία της πρώτερης ε, συνθήκη, δηλαδή να συμμε... υπάρχει συνεργασία Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άκουσα πολλέ παρεμβάσει που είχαν περιεχόμενο υψή του επίπεδου. Έθεσαν σημαντικότατα ζητήματα όσον αφορά το αστικό δίκαιο, όσον αφορά του ανήλικου, όσον αφορά τη μετανάστευση. Εγώ ανέφερα κάποιες προτεραιότητες. Ε, Διερωτώ με, ποια θα είναι η συνέπεια αυτής της συνεισφοράς που πιστεύω ότι έχει αξία. Τι θα συμβεί, τι θα πορεύσει από αυτή τη ε, συζήτηση. Δεν περιμένω άμεσες απαντήσεις. Αλλά αν αυτή είναι μια νέα πορεία, εγώ θα ήθελα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργηθεί ένας οργανισμός, ένας φορέας επεξεργασίας, εμβάθυνσης, που θα εγγυηθεί την ανάπτυξη και προώθηση της συζήτησής μας, να δώσει αποτέλεσμα στη συζήτηση. Αλλιώς θα είναι άλλη μια συνεδρίαση όπου ο καθένας από εμά θα εκφράζει εμπειρίες, θα εκφράζει προσδοκίες, αλλά μετά αυτό δεν θα μεταφραστώ σε κάτι συγκεκριμένο. Εγώ θα ήθελα να αρχίσει να διαγράφεται μια στατηγική που θα δώσει κάποια εγγύηση ότι αυτή η συνεισφορά, αυτή η προσπάθεια δώσει αποτελέσματα. Δηλαδή, οι βουλευτές μέσω των ομάδων και των επιτροπών ε, να ενημερώνονται σχετικά με το τι σκέφτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κάθε επιτροπή του Κοινοβούλιο, ποια είναι η άποψη των επιτροπών και του Κοινοβουλίου για τη συνεισφορά μα, τι συνέχεια θα δώσουμε, ποια στοιχεία θα εξετάζουμε μαζί, ποια στοιχεία θα εξεταστούν σε ένα επίπεδο χαμηλότερο βάσει της κλίμακας αυτών των προτεραιοτήτων και αξιολόγησης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πριν το λόγο στον εισηγητή, θα ήθελα να σχολιάσω κι εγώ Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η δικαιοσύνη, η εφαρμογή του νόμου και η ασφάλεια των πολιτών είναι κάτι που έχουν υπόψη τους ε, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όλη την Ευρώπη και είναι αυτή και η προσδοκία τους. Αυτό περιμένουν από τα κράτη-μέλη σε επίπεδο εθνικό και περιμένουν επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει κάτι αντίστοιχο. Πιστεύω ότι είναι δική μας ευθύνη να βρούμε τρόπους να τα εξασφαλίσουμε όλα αυτά. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμη σίγουρα είναι ένα καλό εργαλείο και θα ήθελα να συνεχίσουμε σε αυτά που είπε ο κ. Μαριτάτη, να συνεχίσω πάνω σε αυτά που είπε και να πω ότι πράγματι χρειάζεται μια δομή η οποία θα είναι σε θέση να αναπτύξει περισσότερο ε, κάποια ζητήματα Ήδη έχω αναφέρει την ΚΟΣΑΚ. Έχουμε 20 χρόνια εμπειρία από την ΚΟΣΑΚ και αυτή η εμπειρία μας δείχνει ότι όταν συζητούμε ζητήματα, όταν, όταν τα συζητούν τα ζητήματα οι διάφορες επιτροπές, όπως οι επιτροπές ευρωπαϊκών υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων στην περίπτωση της ΚΟΣΑΚ, όταν συζητούνται λέγω θέματα από εθνικούς βουλευτές, τότε είμαστε σε θέση να βρούμε κοινό έδαφος, να βρούμε τρόπους για την επίτευξη κοινών στόχων. Και νομίζω ότι αυτός ο τομέας της δικαιοσύνης, της ασφάλειας, ο τομέας της ενόμου τάξεως ε, χρειάζεται πράγματι ε, μια παρόμοια δομή, μόνιμη, όπως είναι η ΚΟΣΑΚ, μια βάση, μια πλατφόρμα και από εκεί να κινούμαστε για ε, κοινή προσέγγιση και συγκεκριμένα βήματα πρέπει να κάνουμε, πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτά ήθελα να πω. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας τώρα, ο οποίος θα συνοψίσει τη συζήτησή μας. Eh, Ευχαριστώ. Ε, αρχικά διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη ομοθυμία σε σχέση με τις φιλοδοξίες κατάργειες του εκτελεστού τίτλου, παρότι υπάρχουν διάφορα εκρεμή ζητήματα που πρέπει να ρυθμίσουμε. Ακούσαμε διαφορετικές απόψεις. Μιλήσαμε για διαφορετικά νομικά συστήματα, διαφορετικό τρόπο λήψης διοικητικών αποφάσεων, ένα κράτος μέλος, αλλά υπάρχει και ένας τρόπος ε, να ενισχύσουμε τη συνεργασία. Γενικά, ξαναλέω, υπάρχει μεγάλη ομοθυμία για αυτό το ζήτημα και ε, ισχυρέ ε, φιλοδοξίε για να, κάνουν, να σημειωθεί πρόοδο. Μιλήσαμε για εναρμόνιση των νομοθεσιών σε διάφορου τομεί του δικαίου οικογενειακό δίκαιο, παραδείγματος χάρη, που είναι ένας ε, τομέας ε, που, όπου μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά προβλήματα σε διασυνοριακέ υποθέσεις. Η κατάργηση του εκτελεστού τίτλου πάντως είναι το αυτονόητο βήμα αν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση ανεξάρτητα αν θα τελεσφορήσει το εγχείρημα ή όχι. Χρειαζόμαστε προσέγγιση των νομικών συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα προσεγγίσουν ναι, και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, των διαφόρων κρατών μελμέντος δε και θα μπορέσουν να γίνουν βήματα προόδου. Τώρα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος για την κατάργηση του εκτελεστού τίτλου, Υπάρχει γενικότερο θέμα ε, και δηλαδή ανάγκη συζήτησης όλων των νομικών ε, ζητημάτων και των διαφορών ε, των εθνικών νομικών παραδόσεων, αλλά με τη συνεχή δουλειά μας επιτυγχάνουμε όλο ένα και μεγαλύτερη προσέγγιση. Ιδού, έτσι μπορώ να συνοψίσω τις συζητήσεις μας, αυτές που κάναμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Θα κάνω κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις, αλλά πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τον κύριο Μέντες Δεβίγκα. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο εισηγητής μας συνόψισε άριστα τη συζήτησή μας και τα όσα υπόθηκαν τα διάφορα στοιχεία αύριο στα συμπεράσματα που θα συνταχθούν απόψε. Ελπίζω στα συμπεράσματα λέγω να μην το παρατραβήξει κυρίως με το καλό κρασί που θα ρέει εδώ στις Βρυξέλλες. Ο συνάδελφος από την Ιταλική Γερουσία αναφέρθηκε σε κάτι που θεωρώ σημαντικό και εγώ. Ίσως θα μπορούσατε συντάξετε τα συμπεράσματα με τέτοιο τρόπο που θα θεσμοθετούνται αυτές οι συναντήσεις. Να μην είναι ακόμα μια συνάντηση αυτή και να έχουμε κρεμί συμπεράσματα χωρίς να δείτε κάποια συνέχεια. Ίσως τα συμπεράσματά σας θα μπορούσατε να προτείνετε να αναβαθμιστούν οι επαφές μας και να θεσμοθετηθούν. Ε, αυτό είναι το βασικό που θέλω να πω έχουμε και παροιμία στη γλώσσα μας. Ότι κάποιος ε, που είναι λακωνικός είναι δύο φορές καλός ρήτορας από κάποιον ο οποίος ε, μακρηγορεί, λέει στη χώρα μας. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Σας ευχαριστώ. Περιμένω σας δω και αύριο επίσης. Σας ευχαριστώ κύριε Μέντες Δεβίγο. Ευχαριστώ κύριε Αυσάν, σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και που συμβάρατε στη συζήτησή μας και υπήρξατε επικοδομητικοί. Να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς, χάρη στους οποίους μπορέσαμε να συνεννοηθούμε. Να υπενθυμίσω ότι το επόμενο, το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας είναι δείπνο που διοργανώνεται από τον πρόεδρο ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Γέρζι Μπούζεκ, στις 7 και 4 το βράδυ, στο εστιατόριο των Ευρωβουλευτών στο κτίριο Henri Spack, Paul Henri Όταν βγείτε, στρίψτε δεξιά και πηγαίνετε στο ισόγειο σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και καλό σας βράδυ. Γεια σας.